Ένωσης και Ρωσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, απαντήσατε σε 38 απαντήσεις. Έχετε ακόμα 5 λεπτά για να πείτε τα τελευταία και καταληκτικά λόγια. Thank you very much. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank, uh, all of you, uh, for... Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις σας Νομίζω ότι από αυτό που ακούστηκε επιβεβαιώθηκε ότι και η Επιτροπή Μεταφορών και η Επιτροπή Ήτρε είναι ιδιαίτερα ισχυρές στην αφοσίωσή τους ε, για την Ευρώπη, στην Ευρώπη και στην προσπάθεια αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Πολλοί από εσά έχετε εργαστεί στα θέματα των μεταφορών εδώ και αρκετό καιρό είσαστε αρκετοί που ήσασταν υπουργοί μεταφορών, κάποιοι μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό, πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ειδικοί στις μεταφορές εδώ και πολλά χρόνια. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι καλό για τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί στον τομέα των μεταφορών τα επόμενα χρόνια, η επόμενη φάση χρονική θα είναι ιδιαίτερος κρίσιμη. Εδώ μπορώ να το συνδέσω αυτό με τις ερωτήσεις τις οποίες ε, μου θέσατε και εσείς. And uh, the future of uh, transport area. Νομίζω ότι εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ε, αυτό που πιστεύω για τον τρόπο με τον οποίο θα κριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μετά από πέντε χρόνια. Απλά κριτήρια καταφέρατε να ανακάμψετε, καταφέρατε να δημιουργήσετε νέες θέσεις απασχόλησης, καταφέρατε να προπαρασκευάσετε την Ευρώπη στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, να την κάνετε πιο ανταγωνιστική. Το κάνατε αυτό με τον ευρωπαϊκό τρόπο, δηλαδή φιλικά προς το περιβάλλον. αιφόρος ανάπτυξη με υψηλά κοινωνικά κριτήρια. Φυσικά αυτές οι ερωτήσεις ε, που θα τεθούν μετά από πέντε χρόνια δεν θα είναι εύκολες ερωτήσεις γιατί κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα είναι κριτής. Πάντως πιστεύω ότι έχουμε τα μέσα για να πετύχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω με τις κοινέ μας προσπάθειες θα το καταφέρουμε. Ξέρετε πολλοί από εσά που έχουμε συνεργαστεί στην προηγούμενη περίοδο ότι είμαι υπέρμαχος της σωστής σχέσης και συντονισμού ανάμεσα στα δύο αυτά κοινοτικά όργανα. Εγώ είχα συνεργαστεί ε, με την διάσκεψη των Προέδρων των, ε, προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τους Προέδρους της Επιτροπής σας δηλαδή και νομίζω ότι θα συνεχίσω προς την κατεύθυνση αυτή μια σωστά ε, διαρθρωμένη στενή συνεργασία. Μένει πάρα πολλά να γίνουν. Η ατζέντα που έχουμε μπροστά μας ε, η κοινή είναι τεράστια. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι τεράστια αλλά νομίζω ότι μπορούμε ε, ε, να το κάνουμε από κοινό και αν με στηρίξετε θα εκμεταλλευτώ τη στήριξή σας αυτή αλλά σε συνεργασία μαζί σας πάντα. Και με αυτή τη δήλωση έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής ακρόασης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλους τους βουλευτές, για τις εμπεριστατωμένες σας ερωτήσεις. Έχουμε καλύψει ένα ευρύ πεδίο της πολιτικής μεταφορών και διαστήματος. Ευχαριστώ και τον υποψήφιο επίτροπο, τον Μάρο Σεύκοβιτς, για τις απαντήσεις που μας έδωσε και για τις θέσεις που πήρε. Υπενθυμίζω στους συντονιστές και τους αντιπρόεδρους της ε, Επιτροπής μας ότι η συνεδρίαση για την ακρο αξιολόγηση της ακρόασης θα γίνει στο α1G2 στις 9.30 και θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω και τους ε, διερμηνείς για τη θαυμάσια εργασία τους και την εγκαρτέρησή τους και τους ευχαριστώ γιατί ξεπεράσαμε λιγάκι και το χρόνο που προβλεπόταν για την ακρόαση. Βλέπετε ότι έχει Πράγματι εκτιμηθεί το έργο σας και σας εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ. Γεια σας.